για την υποστήριξή τους και ευχαριστώ όλους όσοι έλαβαν το λόγο μόνο ότι πολλοί εκφράστηκαν και με, με αντίθετη άποψη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έτσι ολοκληρώθηκε η συζήτηση και αύριο θα γίνει ψηφοφορία. Αγαπητοί συνάδελφοι, το επόμενο θέμα της ημερησίας διατάξεως είναι τώρα η έκθεση της κυρίας Ματιό σχετικά με την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση μίας ενιαίας αδείας διανομής και εργασία στην επικράτεια κράτους μέλους. Και καταρχήν έχει το λόγο η κυρία Ματιό για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Όπως γνωρίζετε, εδώ και 10 χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να αποκτήσει ένα νομοθετικό μέσο σε ζητήματα οικονομικής μετανάστευσης με μια αρχική σφαιρική, σφαιρική προσέγγιση, η Κομισιόν προτίμησε μια κλαδική προσέγγιση. Αυτή η πρόταση οδηγία ε, καταδεικνύει την ανάγκη μια κοινή πολιτική σε θέματα νόμιμη μετανάστευση και δι σε οικονομική μετανάστευση. Μέχρι τώρα νομοθετήσαμε επί θεμάτων παράνομη μετανάστευση, ελέγχου των συνόρων, πολιτική ε, των ε, προξενικών θεωρήσεων. Είναι καιρό να προχωρήσουμε μαζί σε θέματα οικονομική μετανάστευση που η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει και ε, αντιμετωπίζουν όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές οι προκλήσεις είναι η γύρανση του πληθυσμού και το δημογραφικό πρόβλημα. Λόγω αυτών των δύο κακών λοιπόν, που θίγουν την Ευρώπη, τα ζητήματα της ε, ε, τα εργατικά ε, μας αναδεικνύουν τις ελλείψεις που υπάρχουν. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται να βρεθούν λύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να επιλύσουμε το πρόβλημα και η οικονομική μετανάστευση είναι, μια, είναι ένα θέμα που χρειάζεται να μας απασχολήσει και να ε, διερευνήσουμε. Δεν έχει όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τις ανάγκες αλλά και τις δυνατότητες υποδοχή κάθε κράτου μέλου. Όπω αναφέρεται στα άρθρα 1 και έω 8 την πρόταση οδηγία, τα κράτη-μέλη είναι κύριοι του όγκου των μεταναστών που μπορούν να δεχθούν στον επικράτειά του. Οι κυβερνήσει θα δρουν με τρόπο διαφορετικό για να ε, υλοποιήσουν την οικονομική μετανάστευση. Διάφορα ρυθμιστικά μέτρα, αλλά μέχρι τώρα κάνουν αυτό το μέτρο, δεν, αυτό το μέτρο δεν μπόρεσε αποτελεσματικά να επιλύσει τα παράνομε μεταναστεύσει, την παράληψη συγγνώμη μεταναστεύσεις. Ε, σχέση μεταξύ τη οικονομική μεταναστεύσης και τη παράτυπης είναι προφανή. Χρειάζεται λοιπόν μόνο με, με συνδυασμένη αντιμετώπιση μπορούμε να επιλύσουμε το πρόβλημα. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχουν αυτά τα μέτρα τα οποία έχει προτείνει εδώ και πέντε χρόνια η Κομισιόν. Τι θα προσφέρει αυτή η νέα οδηγία για την Ενία διαδικασία αίτηση για τη χορήγηση άδεια εργασία για διαμονή με, διαφορά, σε διαφορά με την, κάρτα, με την μπλε κάρτα δεν αφορά την, ε, την ε, άφηξη ε, υπηκών χωρών, αλλά έχει ως στόχο να λιάνει τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στα κράτη-μέλη, προκειμένου τα δικαιώματα να είναι ισότιμα για τους εργαζόμενους που Δεν υπάρχει ακόμα ένα ευρωπαϊκό μέσο για να προσφέρει στους εργαζόμενους τρίτων χωρών που διαμένουν και εργάζονται νομίμως στην Ευρώπη. Αυτή η οδηγία λοιπόν θα μπορέσει να ρυθμίσει αυτές τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στους εργαζόμενους εφαρμόζοντας μια ίση μεταχείριση ανάμεσα στους εργαζόμενους, συνθήκες εργασίας, επαγγελματική κατάρτιση, εκπαίδευση, κοινωνική προστασία, πρόσβαση στις υπηρεσίες και φορολογικά ωφέλη. Μια τέτοια πρόταση θα προσφέρει την ε, εγγύηση της μη εκμετάλλευσης αυτών των ε, προσώπων. Επιτρέπει επίσης την καταπολέμηση του αθέμητου ανταγωνισμού που εφαρμόζεται εις βάρον των Ευρωπαίων εργαζομένων. Αυτό λοιπόν το δίκτυο προστασία θα έχει ως αποτέλεσμα έχει μάλλον ως αποτέλεσμα να ε, προσλαμβάνονται εργαζόμενοι με ελάχιστες ασφάλειες ε, και σε χειρότερες συνθήκες εργασίας. Όλα τα κρατη λοιπόν θα έχουν μια τυποποιημένη ε, διαδικασία πολύ πιο γρήγορη στην εφαρμογή της. Ε, θέση αυτής της οδηγίας θα προσφέρει πλεονεκτήματα στους μετανάστες, στις διοικήσεις, στου εργοδοτές και θα επιτρέψει με καλύτερη διαχείριση των νόμιμων μεταναστευτικών δρόμων. Το Κοινοβούλιο σήμερα είναι εσύ κάτι το οποίο σημαίνει ότι χρειάζεται να δείξει την απαραίτητη υπευθυνότητα. Πρέπει λοιπόν να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων που μας προσφέρει η συνθήκη της Λισαβόνας. Ας είμαστε λοιπόν αξιόπιστοι συνομιλητές και να μπορέσουμε να επιλύσουμε αυτή την πρόκληση που χτυπάει τις πόρτες της Ευρώπης. Νομίζω ότι μια τέτοια οδηγία θα είναι υποφελής για όλους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την Επιτροπή και πάλι Επίτροπος Μάλστρομ. Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Ματιό και τον κύριο Θέρκα στους δύο συγητές και τις δύο επιτροπές όπως επίσης και την Βελική Προεδρία για την πολύ ε, σκληρή δουλειά που έκαναν. Όπως είπε και η συγητρία, η Κομισιόν υπέβαλε αυτή την έκθεση το 2007 ο στόχο ήταν και είναι η απλοποίηση των διαδικασιών με την εισαγωγή μιας άδεια εργασίας και διαμονής, ενώ παράλληλα θα εγγυόμαστε τα δικαιώματα εργασία ε, στου ε, νομίμως ε, διαμένοντε σε χώρες Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν καλύπτονται από άλλα νομιστικά κείμενα. Δεν συζητούμε για τους όρους χορήγησης ή απόρριψης ε, αιτήσεων. Αυτή, αυτοί οι όροι εμπίπτουν στις ε, εθνικές αρμοδιότητες καθώς επίσης και στα αριθμητικά όρια αν υπάρχουν. Ε, η, η πρότασή μας όμως ε, αποτελεί ακρογωνίο λίθο της ευρωπαϊκής ε, πολιτικής εργασιακής ε, μετανάστευσης. Αν εγκριθεί θα γίνει σαφής η προσφορά των επικών αυτών τρίτων χωρών στις χώρες μας. Η πρόταση είναι περίπλοκη, πολύ περίπλοκη. Υπάρχει μια μεταναστευτική πλευρά και μια πλευρά εργασιακή κοινωνική. Η πλειοψηφία των ε, τροπολογιών που ψηφίστηκαν από τις Επιτροπές ε, υποστηρίζονται από την Κομισιόν διότι ενισχύουν τις ε, εγγύησεις, τις διαδικαστικές εγγύησεις και για τους εργαδότες και για τους εργαζόμενους. Για παράδειγμα, τροπολογίες για την περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών και ενίσχυση των διατάξεων ίσης μεταχείρισης με την, την ρήτρα αναλογικότητας των τελών κλπ, φορολογικών κινήτρων κλπ. Απ' την άλλη μεριά, ε, προαπαιτείται ε, η ύπαρξη διμερής συμφωνία για τη μεταφορά συνταξιδοτικών δικαιωμάτων, κάτι που είναι πιο ε, αυστηρό από αυτό προτείνει η Κομισιόν. Ε, βλέπω ότι το Κοινοβούλιο έκανε προσπάθεια συντονισμού των θέσεων των ε, ε, ε, πολιτικών ομάδων. Θα κάνουμε και εμείς προσπάθεια. Ξέρουμε ότι έχετε λάβει υπόψη επίσης πολλές, πολλά αιτήματα του, του Συμβουλίου. Ε, θα πρέπει να γίνουν σεβαστά διάφορα κριτήρια όπως ο στόχος καθώς επίσης και η ανάγκη χορήγησης ενιαίων δικαιωμάτων από την έναρξη της εργασίας τους στις χώρες μας. Επίση, χρειάζεται ε, μια ενιαία αντιμετώπιση όλων αυτών των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι σημαντικό να δείξουμε στου εταίρου μα ότι ε, θέλουμε να εξασφαλίσουμε την ε, δίκαιη μεταχείριση των υπηκών τρίτων χωρών που εργάζονται και διαμένουν νόμιμα στις χώρε μα. Ε, υπάρχουν βέβαια δημοσιονομικά θέματα σε ό,τι αφορά την ίση μεταχείριση, αλλά είμαι σίγουρος θα τηρηθούν και τα δύο προηγούμενα κριτήρια παρόλο ότι η, πρόταση, η τελική πρόταση δεν είναι τόσο αισιόδοξη όσο η αρχική, όσο περιμέναμε. Είναι μια καλή πρόταση παρόλα αυτά. Είναι ένα σημαντικό βήμα στον τομέα τη νόμη μετανάστευση. Πιστεύω ότι θα είναι πολύ σημαντική για του εργαζόμενου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζω λοιπόν ότι θα καταλήξουμε συμφωνία σε, αυτή την, σε αυτό το κείμενο το σύντομα το δυνατό. Ευχαριστώ ξανά τους ηγητές και τους σκιώδεις ηγητές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Επίτροπε και τώρα για την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ο κύριος Τσέρκας για τέσσερα λεπτά. Καλησπέρα κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Η μετανάστευση στην Ευρώπη είναι ένα γεγονός πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό πρόορης της ε, σημασίας αποτελεί μια τεράστια ευκαιρία, αλλά χρειάζεται παράλληλα μια ευθύη διαχείριση και δίκαιη. Διαφορετικά θα αποτελέσει πρόβλημα και ε, δεν θα έχουμε αντιμετωπίσει με τρόπο δίκαιο τους εργαζόμενους οι οποίοι ε, θα απειληθούν, ε, χάσουν την θέση τους κλπ. Και θα έχει ως αποτέλεσμα έναν διχασμό του εργασιακού χώρου και καταστροφή του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου. Γι' αυτό λοιπόν κύριε Επίτροπε η, ισότιμη μεταχείριση είναι η κλίδα για την επίλυση του προβλήματο με τρόπο δικαίο και ευφύ. Το Συμβούλιο το είπε και στο Τάμπερ προετών. Η Κομισιόν το είπε πριν από πέντε στην Πράσινη Βίβλο και το Κοινοβούλιο αύριο θα αποφανθεί επί μιας προτάσεως για μια νομοθετική πρόταση. Και το τρίτο κεφάλαιο τη Οδηγία δεν είναι μονογραφειοκρατική αλλά είναι μια οδηγία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που θα πρέπει να εφαρμόζονται σε όλους ε, τους ε, μετανάστες ε, προκειμένου να την χάνουν ισόρυμες μεταχείρισης. Δυστυχώς όμως η οδηγία δεν είναι αυτή την οποία μας είχατε αναγγείλει και το λέω εγώ, το λέει η Επιτροπή Επασχόλησης διότι όλες και επίση όλες οι μη κυβερνητικές οργανώσεις που ασχολούνται με το θέμα, όλες οι εκκλησίες και όλες τα συνδικάτα. Αυτή η οδηγία λοιπόν είναι ανεπαρκής και είναι και επικίνδυνη για δύο λόγους. Πρώτον, διότι αποκλείει τους, ε, αυτούς που έχουν, ε, έχουν ανάγκη από στήριξη, τους, ε, τα άτομα τα οποία έχουν έρθει ως πρόσφυγες και άλλους θα εφαρμοστεί η αρχή της χώρας καταγωγής νομίζω επίσης ότι τα άτομα αυτά θα πρέπει να καλύπτονται όπω είπε η κυρία Ματιέ αλλά εσεί με την οδηγία επιτρέπετε ακόμη στα άτομα τα οποία καλύπτονται να αφήνετε η δυνατότητα να εξαιρούνται από την ίση μεταχείριση σε ό,τι αφορά την <clears throat> τη συνταξιοδότησή του, τον επιστρέφουν τη χώρα του, τα κοινωνικά προνόμια τα οποία θα ε, μπορούσαν να έχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση, αποκλείονται από τις υποτροφίες κάθε είδους στήριξης για την επαγγελματική του εκπαίδευση και κατάρτιση. Η Κομισιόν ε, στα σκεπτικό αναφέρει τον αντίκτυπο ε, μελέτη, τον μελέτη και ότι θα πρέπει να καταργηθούν ε, οι διακρίσεις, αλλά στην ουσία αυτό δεν συμβαίνει κύριε Επίτροπε. Επίσης έχουμε και τροπολογίες που έχουν παρουσιάσει οι ομάδες της δεξιάς και της κεντροδεξιάς που πάνε ακόμα παραπέρα. Παίρνουν ε, θέσεις πολύ πιο ακραίες από το Κοινοβούλιο για να καταστρέψουν την ε, ομοφωνία που πετύχει, τη συνέντευξη μάλλον που πετύχαμε στην Επιτροπή Αποσχόληση. Νομίζω λοιπόν, συνάδελφοι, ότι χρειάζεται να κάνουμε μια ζήτηση πολύ ευρύτερη μεταξύ μα επί του θέματο σε σχέση με τι άλλε οδηγίε να είμαστε ανοιχτοί στι ε, κοινωνία της Ευρώπης, στις ε, μη κυβερνικές οργανώσεις, στις εκκλησίες, να μην βιαστούμε λοιπόν, να μην το αντιμετωπίσουμε στα βιαστικά στο πόδι, εγκρίνοντας αύριο το κείμενο του Συμβουλίου. Νομίζω λοιπόν πως η πλειοψηφία των συναδέλφων θα συμφωνούσαν το να κάνουμε μια ευρύτατη συζήτηση για να πετύχουμε ευρύτατη συνένεση στο Κοινοβούλιο που θα σέβεται τις αρχές των, ε, της Χάρτας Δικαιωμάτων που θα δέχεται τις ε, συστάσεις ε, της ε, Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας είναι κάτι το οποίο αφορά την μέλλον της Ευρώπης. Στην Ευρώπη χρειαζόμαστε όλοι οι εργαζόμενοι, χωρίς καμία εξαίρεση, όποια και αν είναι η χώρα καταγωγής, να έχουν όλα τα δικαιώματα. Με αυτός είναι ο τρόπος για να καταπολεμήσουμε το ρατσισμό και την ξενοφοβία για μια Ευρώπη δίκαιη και αξιοπρεπή. Ευχαριστώ. Τώρα ερχόμαστε στους ομιλητές εν των πολιτικών ομάδων και για το ΕΛΚ μιλάει η κυρία Όμαν Ρόιτερ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να συγχαρώ καταρχήν την κυρία Ματιό γιατί ε, ανάλαβε ένα θέμα το οποίο χρονολογείται από παλιά. Κυρία Μάλστρομ, το 2001 υποβλήθηκε μια, ένα προσχέδιο πρότασης για τους ε, όρους που επιβάλλονται σε επικόστη των χωρών για την ασύγκριτη και τη διαμονή τους. Ε, αυτή η πρόταση αποσύρθηκε το 2006 και ε, υποβλήθηκε μια καινούργια πρόταση για μια ενιαία διαδικασία ε, υποβολής αίτηση για άδεια διαμονής και εργασία μαζί. Εγώ έτσι και έχω καταλάβει το ιστορικό. Δεν συμφωνώ πλήρω με τον κύριο Θέρκας οι υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν μία ενιαία άδεια θα έχουν κοινωνικά δικαιώματα. Τα κοινωνικά δικαιώματα όμω πρέπει να καλύπτουν του πάντε. Αυτό είναι αλήθεια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Θέρκα γιατί πάντοτε είναι ευχάριστο να μιλάω μαζί του. Το συζητήσαμε στην Επιτροπή ε, Κοινωνικών Υποθέσεων και συζητήσαμε ακριβώ το θέμα του πεδίου εφαρμογή. Ε, αποσπασμένοι εργαζόμενοι δεν ε, είναι δυνατόν να ε, χαίρουν τέτοιου καθεστώτος ενίας ε, διαμονής και εργασίας. Στην αντίστοιχη οδηγία απόσπασης υπάρχουν άρθρα τα οποία έχουν σχέση με αυτό το θέμα και πιστεύω ότι τα δικαιώματα τους έχουν ήδη τύχει επαρκών εγγύσεων σε εκείνη την οδηγία. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι, τρί, οι υπήκοοι τρίτων χωρών δεν θα προσφέρουν τις ε, υπηρεσίες τους με χειρότερους όρους από ότι οι εθνικοί υπήκοοι. Ένα άλλο θέμα <clears throat> ε, για το οποίο είχα πρόβλημα ήταν το θέμα της ίσης μεταχείρισης. Είχα υποβάλει τροπολογία και έγινε δεκτή. Ο κανονισμός 883 προβλέπει το θέμα της ε, ε, ίσης μεταχείρισης, προβλέπει την ίση μεταχείριση ε, και χαίρομαι που ο συμβασμός ήταν θετικός τελικά, επετεύχθη γιατί η ίση μεταχείριση πλέον την χάνει επαρκών εγγύσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τώρα για τους σοσιαλιστές η κυρία Μπλικεβιτσούδε για τρία λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ με συγχωρείτε αλλά δεν υπάρχει διερμηνία σε όλε τι γλώσσε, λέει η πρόεδρος ρωτάει η, η ομιλήτρια υπάρχει τώρα διερμηνία ευχαριστώ για προχωρήστε τώρα Κυρία Επίτροπε, κυρία Ματιά, αγαπητοί συνάδελφοι, όντως αυτή η οδηγία που αναφέρεται εις ε, την ενιαία άδεια διαρμονής και εργασίας είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση η οποία χρειάστηκε πολλή συζήτηση και εξεφράστησαν πολλές γνώμες αλλά δεν μπόρεσε να υπάρξει μια ενιαία αποδοχή για τους ε, εργαζόμενους από όλες τις τρίτες χώρες που εργάζονται νομίμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επρόκειτο για ένα πλαίσιο οδηγίας που θα αποτελέσει τη βάση για εξειδικευμένες οδηγίες διότι μόνο έτσι θα μπορέσει κανείς να υλοποιήσει τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως να υπάρξει μία ενιαία ε, μεταναστευτική πολιτική. Αλλά η νομική βάση την οποία μας είχαν υποσχεθεί εξαφανίστηκε εφόσον ε, δεν θα εφαρμόζεται ε, αυτό το σύστημα σε ορισμένους εργαζόμενους όπως οι εποχιακοί αποσπασμένοι πρόσφυγες και αυτοαπασχολούμενοι. Άρα δεν θα μπορέσει να καλύψει όλους τους εργαζόμενους και θα αποτελέσει μόνο ένα σημείο αναφοράς και θα χρειαστεί να διευρύνουμε την εφαρμογή της σε, όλους τους, σε όλες τις κατηγορίες εργαζομένων και ιδίως στους εποχιακούς διότι διαφορετικά δεν θα μπορέσει να υπάρχει δικαιοσύνη και ισότητα στην, εργασία, στην αγορά εργασίας. Θέλω να τονίσω ότι οι νόμιμοι μετανάστες συμβάλλουν στην οικονομία των χωρών όχι μόνο μέσω της εργασίας τους αλλά και μέσω της φορολογίας και των κοινωνικών εισφορών. Πρέπει λοιπόν να χαίρουν των ίδιων δικαιωμάτων και να χαίρουν μία ε, ίση μεταχείρισης στην αγορά εργασίας. Αύριο πρέπει να είμαστε συσπηρωμένοι για να ε, πετύχουμε σε αυτή τη μάχη, δηλαδή όλοι να, όλοι οι εργαζόμενοι να χαίρουν των ίδιων δικαιωμάτων βάσει της εφαρμογής αυτής της οδηγίας. Δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε μία αγορά εργασίας δύο ταχυτήτων, δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε μία τάξη εργαζομένων δευτέρας κατηγορίας χωρίς δικαιώματα και χωρίς εγγυήσεις, διότι τότε όλα τα κεκτημένα μας θα είχαν καταπο... καταπατηθεί. Ευχαριστώ και τώρα η κυρία Ίνφελτ για δύο λεπτά εν ονόματι των φιλελευθέρων. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ξεκινήσω με ένα διαδικαστικό, διότι βλέπω ότι για μία τόσο σημαντική συζήτηση ο ομόλογός μας στο Συμβούλιο δεν ε, παρίσταται και το βρίσκω απαράδεκτο διότι θα και σκοπεύω να γράψω στο Συμβούλιο και να παραπονεθώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θα ε, ήθελα όμως καταρχήν να συγχαρώ την κυρία Ματιό που έκανε εξαιρετική εργασία σε ένα πολύ δύσκολο και πολύ ευαίσθητο θέμα που ε, εξετάζει αυτός ο Φάικελος διότι και η δικιά μας πολιτική ομάδα θέλει να καταλήξει σε μία συμφωνία διότι αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πολύ σημαντική αυτό όμως χωρίς μεγάλη ευχαρίστηση γιατί όπως έχει εκφραστεί με διαφορετικά λόγια λόγια από οι προλαλήσαντες και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύουμε ότι η πρόταση αυτή δεν προχωρά όσο προοδευτικά θα έπρεπε και όσο χρειάζεται. Χρειάζονται επίση και επιπλέον έγγραφα. Δηλαδή αν, ζητήσουν, αν μπορούν τα κράτη να ζητούν επιπρόσθετα έγγραφα τότε αλλήμονό μα Δεν, ε, δεν εξυπηρετεί το στόχος. Με την ενιαία άδεια δεν χρειάζεστε άλλα έγγραφα. Θα ήθελα δε να σας πω ότι για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία η πολιτική μου ομάδα δεν ε, ε, θα ε, δεν θα υπερψηφίσει τους πίνακες συσχετισμών και θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο μέρος των κρατών μελών διότι εάν τα κράτη-μέλη ήταν διάφανα θα έπρεπε οικειοθελώς ε, να περιλάβουν τους πίνακες συσχετισμού. Και τέλος θέλω να σας πω, το 1999 στο Τάμπερε είχαν ε, διακηρύξει τα κράτη-μέλη ότι θέλουν μια κοινή μεταναστευτική πολιτική. Μέχρι σήμερα πόσο έχουμε προδοθεί εκπαιδεύσει σχεδόν καθόλου. Τα κράτη-μέλη δεν θέλουν μια κοινή μεσαναστευτική πολιτική. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τώρα για την ομάδα των Πρασίνων ο κύριος Λάμπερτ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και μας, μας ε, ανησυχούν οι διαφορές ε, στην ε, αγορά μεταξύ των 27 κρατών ε, μελών οι ε, διαφορές στα ρεσιακά δικαιώματα κλπ. Το θέμα είναι όμως πώς μπορούμε να πάμε σε μια πιο ισχυρή κατάσταση ε, και πιο ενιαία κατάσταση. Ε, είναι σίγουρο ότι χρειάζονται κοινά δικαιώματα για τους υπηκόους τρίτων χωρών όπως τα είχε προτείνει αρχικά η Κομισιόν και βελτιώθηκαν από την Επιτροπή Απασχόλησης. Δεν θέλουμε αυτά τα δικαιώματα να περιορίζονται και να περικόπτονται διαρκώς. Θα υποστηρίξουμε αύριο την, ε, τα, την πιο ευρία γκάμα δικαιωμάτων ε, είναι, είναι δυνατή. Ε, τα, οι πολίτες τρίτων χωρών θα πρέπει επίσης να χαίρουν τη δυνατότητα ε, εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς επίσης και μεταφράση δεξιδοτικών δικαιωμάτων όπως είχε αναγνωριστεί και στην ε, πρόταση ε, η εργασία τους βοηθάει και την κοινωνία μας αλλά πρέπει να χαίρουν αυτών των δικαιωμάτων επίσης το θέμα της ε, κυκλικής μετανάστευσης είναι πολύ σημαντικό το πεδίο εφαρμογή είναι επίμαχο θέμα διότι υπάρχουν και άλλα νομιστικά κείμενα τα οποία συζητώνται αυτή τη στιγμή ή υπάρχουν δεν θα πρέπει να αυταπατώμεθα ότι αυτό το κείμενο το οποίο συζητούμε μπορεί να καλύψει όλους τους εργαζόμενους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειαζόμαστε ε, μια πιο προσαρμοσμένη προσέγγιση έτσι ώστε η μετανάστευση να λειτουργεί για όλους. Ε, δεν θα υπερψηφίσουμε την συμπερίληψη ανθρωπιστικών δικαιωμάτων για παράδειγμα. Για την Ηνωμένη Αριστερά, ο κύριος Λεαρίκ για δύο λεπτά. Κυρία Πρόεδρε, Κύριε Επίτροπε, όπως ε, παρατήρησε πολύ σωστά ο κύριος Σέρκας, υπάρχει διαφωνία ανάμεσα στην Επιτροπή Απασχόλησης ε, και ε, ελευθεριών. Το κοινοβουλίο μας λοιπόν θα πρέπει να αρνηθεί να εγκρίνει αυτή την οδηγία για την ενιαία άδεια. Αυτός, αυτή η οδηγία έχει μόνο ένα στόχο, δηλαδή να θέσει τους Ευρωπαίους εργαζόμενους σε ανταγωνισμό σε σχέση με τους εργαζόμενους εκτός Ευρώπης αλλά και ανάμεσα στους μετανάστες εργαζόμενους. Εάν η οδηγία παραμείνει ως έχει θα έχουμε διάφορα καθεστώτα των διαμενόντων, των ε, ε, μεταντιθεμένων ενδοπιχειρησιακά, των εποχιακών κλπ. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε πολλές κατηγορίες εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό θα παραβιάζει τις αρχές της χάρτας ε, των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αντίθετα από το που είπατε κυρία εισηγήτρια, με τέτοιες διαφορές καθεστώτων αυτό θα οδηγήσει σε μια μόνιμη υποβάθμιση των συνθήκων εργασία όλων των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ισότητα δεν μπορεί να περιοριστεί μόνο στην αναφορά των συνθήκων εργασία. Όπω είπε ο κύριο Έρκα, η ισότητα χρειάζεται να αφορά του μισθού, τι αμοιβέ, τον χρόνο εργασία, την υγεία, την ε, κοινωνική προστασία, την πρόσβαση στι δημόσιε υπηρεσίε, την κατάρτιση. Εάν δίχως αυτόν τουλάχιστον παρονομιστεί, τότε θα έχουμε μια ζούγκλα ε, ε, και μια συνεχής εκμετάλλευση. Η ισότητα χρειάζεται να αφορά όλους τους ε, εργαζόμενους και εργαζόμενες όποια και αν είναι η καταγωγή τους. Δεν θα πρέπει να προσθέσουμε νέους ανταγωνισμούς ανάμεσα στους εργαζομένους ε, επιπλέον της απαράδεκτης οδηγίας Μπολκενστάιν. Θα πρέπει λοιπόν να τονίσουμε την αρχή της ε, ισότητας ε, διαφορετικά δεν θα πετύχουμε την κοινωνική Ευρώπη, την ουμανιστική Ευρώπη κάτι το οποίο ε, θα πρέπει να μας οδηγήσει να απορρίψουμε αυτή την οδηγία. Ευχαριστώ. Και τώρα για την Ένωση Ελευθερίας και Δημοκρατίας ο κύριος Μπιζότο για ένα λεπτό. Η κυρία Μπιζότο. Αγαπητοί συνάδελφοι, η προσυζήτηση οδηγία περιέχει διάφορα θετικά στοιχεία. Ε, το γενικότερο ζήτημα είναι η υπέρβαση κάποιων γραφειοκρατικών δυσκολιών για του εργαζόμενου τρίνων χωρών και για την ε, ενιαία άδεια Διαμονή και εργασία. Δεν ήθελα να επενθυμίσω όμω πω σήμερα στην Ευρώπη δεκάδες εκατομμύρια πολιτών, μεταξύ των οποίων πολλοί νέοι, είναι άνεργοι λόγω των διαχρονικών ελλείψεων του παραγωγικού συστήματος της Ευρώπης, λόγω μιας κρίσης η οποία φαίνεται ότι δεν τελειώνει ποτέ. Ε, πρώτα από, εκτός από τους πολίτες τρίνων χωρών που διαμένουν στις χώρες μας, η Ευρώπη θα πρέπει να επιτρέψει τη λήψη νέων πολιτικών και κοινωνικών μέτρων, τα οποία θα βοηθήσουν καταρχήν τους πολίτες μας στο να βρουν ή στο να επαναεύρουν εργασία. Εάν η Ευρώπη μπορέσει να δώσει εργασία στους πολίτες της, τώρα θα δημιουργήσει τα τις βάσεις για να μπορέσει να υποδεχθεί τις μεταναστευτικές ροές το σύστημά μας θα πρέπει να είναι να οικοδομήσουμε μια Ευρώπη η οποία θα μπορεί να στέκεται όρθια στα πόδια της και έτσι θα μπορέσουμε να δώσουμε ε, εργασία και στους άλλους. Με συγχωρείτε δυστυχώς τέλειωσε η ώρα σας και τώρα για τους ε, μη εγγεγραμμένους ο κύριος Βάντερ Στόπ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το κόμμα μου ανέκαθεν υποστήριζε πως ε, είμαστε κατά της ε, ευρωπαϊκής πολιτικής ε, στα θέματα τα έχουμε μια εξαιρετική κυβέρνηση στην κάτω χώρες που θα μπορέσει επιτέλους να εφαρμόσει τη βούληση του Ολλανδικού λαού. Αλλά ε, ε, ε, βρισκόμαστε ενώπιον ενός τεταλισμένου γεγονότος. Θα πρέπει αυτές οι αρμοδιότητες να αποδοθούν στα κράτη-μέλη. Εν τω μεταξύ θα πρέπει να περιορίσουμε την καταστροφή. Αλλά αυτό δεν περιέχεται, μπορούμε να το μέσω της οδηγίας. Αυτή η οδηγία φέρνει το αντίθετο αποτέλεσμα. Μόνο μια, μια ελιτίστικη πολιτική τάξη θα επιθυμεί να ενεργήσει. Εγώ εξελέγην από Ολλανδούς ε, πολίτες και από πρόσωπα τα οποία έρχονται να εργαστούν στην Ολλανδία αλλά που δυστυχώς δεν τηρούν τις χριστιανικές αρχές. Εγώ θα την καταψηφίσω την έκθεση. Τώρα ερχόμαστε στους επόμενους εγγεγραμμένους ομιλητές. Πρώτα ο κύριος Μπουσουτήλ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ την Βερονίκ Ματιού για την εξαιρετική εργασία της και για το εξαιρετικό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Θα ήθελα να πω επίσης ότι από πλευράς του ΕΛΚ χρειάζεται να συνεργαστούμε στον τομέα της νόμιμης μετανάστευσης και αυτό και πρέπει να καθιστήσουμε σαφέ ότι καταπολεμάμε την παράνομη μετανάστευση, την λάθρο μετανάστευση. Ταυτόχρονα αναγνωρίζουμε το γεγονό ότι ένα από τα εργαλεία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να πλήξουμε την παράνομη μετανάστευση είναι να ε, προωθήσουμε την ύπαρξη σαφών και ε, καλών ευκαιριών για την ε, νόμιμη μετανάστευση. Να σας υπενθυμίσω επίσης, όπως είπε και η Βερονίκ Ματιέ, ότι η συνθήκη της Λισαβόνας μας δίνει νέες εξουσίες σε αυτόν τον τομέα και νέες ευθύνες. Επίσης, χρειάζεται να είμαστε υπεύθυνοι και να μπορέσουμε να πετύχουμε κάποιου συμβασμού όπου είναι απαραίτητη με το Συμβούλιο των Υπουργών. Χρειάζεται λοιπόν να δεχτούμε κάποιε θέσει του Συμβουλίου, όπω ε, αυτό την προστασία που θέλει να διατηρήσει το Συμβούλιο κατά την ε, έκδοση αυτών των αδειών. Εδώ υπάρχει επίση το ζήτημα τη ίση μεταχείρισης. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε κάποιου συμβασμού για να μπορέσουμε να επιτύχουμε συμφωνία με τον Συμβούλιο. Να καταλήγοντας να πω πως ε, όσοι πιστεύουν ότι βιαζόμαστε ή ότι πρέπει να καταψηφίσουμε θα πρέπει να γνωρίζουν ότι δίχως ε, αυτήν την οδηγία δεν θα μπορέσουμε να δώσουμε να πρέπει αξιοπρέπεια στους εργαζόμενους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τώρα ο κύριος Μωράης για τρία λεπτά. Ε, Όλο και επιμικίνεται το χρόνο ε, ομιλία μου. Θα προσπαθήσω να γεμίσω αυτά τα τρία λεπτά. Ε, οι προηγούμενοι ομιλητέ των σοσιαλιστών ε, εξέφρασαν τα, τα βασικά προβλήματα της ομάδας μας για αυτό το πακέτο. Ε, δεν αφορά μόνο το, το καθεστώς της χώρας προέλευσης ή την ίση μεταχείριση η κυρία Ρόιτε το ανέλησε αυτό, αλλά είναι και θέμα του το, πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Έχουμε μια πρόταση νέα εισόδου ε, που υποβάλλεται μετά την πρόταση για την μπλε κάρτα και μετά τις κυρώσεις ε, για τους εργοδότες. Υπάρχει δηλαδή ένα πακέτο το οποίο είχε μια καλή πρόθεση οριζόντιας προ, προσέγγισης, αλλά τελικά η προσέγγιση δεν είναι οριζόντια. Γιατί ε, κατάσταση είναι εξή. Η κυρία Ματιό κάνει ό,τι μπορεί με αυτό που έχει στα χέρια τη, αλλά το είπε και η ίδια. Θέλαμε μια συνολική προσέγγιση, αλλά τελικά έχουμε τομεακή προσέγγιση. Αυτή η τομεακή προσέγγιση ε, είναι αυτό που ανησυχεί και την κυρία Λάμπερτ. Λοιπόν, πού βρισκόμαστε σήμερα. Ε, εμείς στην ομάδα μας ανησυχούμε ε, σε ό,τι φορά την αρχή της χώρας προέλευσης και όπως είπε η κυρία Μπλινκοβιτσιούτε έχουμε ένα πραγματικό πρόβλημα με τις κατηγορίες των εργαζόμενων που περιλαμβάνονται στην πρόταση. Οι ενδοεπιχειρησιακές μετα... με... ξερούνται και άλλες πολλές κατηγορίες εργαζομένων. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Αν έχουμε μια ενιαία <laughs> άδεια που δεν είναι αυτό που λέει που δεν έχει μια ε, αρκετά επαρκώς ευρία βάση θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα στην ίση μετακίνηση, θα δημιουργήσουμε εργαζομένους δύο ταχυτήτων, δύο επιπέδων ε, που ε, δεν θα μπορούμε να λύσουμε. Από την άλλη μεριά αναγνωρίζουμε και χαιρόμαστε ε, για το γεγονός ότι χρειάζονται, για το ότι έχουμε και τομιακές ε, ρυθμίσεις αλλά εμείς ως ομάδα θέλουμε μια οριζόντια προσέγγιση. Τι να κάνουμε, λέμε την αλήθεια. Κάνουμε τα πράγματα ανάποδα. Γιατί, γιατί κάποιοι οποίοι δεν είναι παρόντες σήμερα, το Συμβούλιο δηλαδή, δεν ήθελαν να ρυθμίσουν το θέμα οριζόντια. Τελικά μείναμε με αυτή την κατακαιρματισμένη προσέγγιση. Αυτή η ενιαία λοιπόν έχει καλές προθέσεις. Αναγνωρίζουμε τις προσπάθειε της ηγετρίας, αλλά θα υποβάλουμε τροπολογίες αύριο καλόπιστα, ελπίζοντας ότι η ενιαία άδεια θα, θα είναι πραγματικά ενία και θα καλύπτει μια ευρεία βάση ε, ανθρώπων, εργαζομένων που θα εργάζονται και θα διαμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα έχουν τα ίδια δικαιώματα και που θα αντέξει το χρόνο. Ευχαριστώ και τώρα η κυρία Μάιστερ για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρέπει να σας πω ότι εδώ και ένα χρόνο είμαι στο Κοινοβούλιο, έχω ασχοληθώ με διάφορα θέματα, αλλά κανένα δεν ήταν τόσο δύσκολο όσο αυτό. Και θέλω να ευχαριστήσω θερμά την κυρία Ματιού και τον κύριο Σέρκα, στους δύο εισηγητές από τις δύο επιτροπές. Ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα, διότι καταρχήν έχουμε υψηλά ιδεώδη στην Ευρώπη. Θέλουμε όλοι να τη χάνουν ίδιας μεταχείρισης στην Ευρώπη και από αυτού συμφωνούμε όλοι το θέμα είναι ε, τι μπορούμε στην πραγματικότητα να υλοποιήσουμε και με την συνθήκη της Λισαβόνης ε, θέλουμε να έχουμε μια κοινή πολιτική ασύλου και μετανάστευσης και η πολιτική της ε, μετανάστευσης είναι κάτι που χρειαζόμαστε διότι έχουμε δημογραφικές αλλαγές και χρειαζόμαστε όχι πολύ κατηρτισμένους αλλά και όχι κατηρτισμένους εργαζόμενους εδώ εδώ. Ε, όπως είπε και η κυρία Έντφελτ, ήδη από το 99 στο Τάμπερ είχαν πει οι αρχηγοί κρατών ότι θέλουμε να κάνουμε κάτι ε, όλοι μαζί. Μέχρι στιγμής όμως δεν έχουμε τίποτα προς Υπάρχει μια συμβιβαστική λύση η οποία δεν μα ικανοποιεί πλήρω, αλλά ήδη ε, συμβιβασμό σημαίνει κάτι που μπορούμε να προωθήσουμε κατά τη γνώμη μου. Χρειαζόμαστε βέβαια χρόνο να συζητήσουμε. Δεν μ' αρέσουν όλα και ιδιαίτερο θεωρώ είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι όλοι πρέπει να έχουν τη δυνατότητα εκπαιδεύσεως και επιμορφώσεως γιατί έχει σημασία όχι μόνο για τους ε, ανθρώπους να είναι ε, κατηρτισμένοι στην αγορά αλλά και εμείς να έχουμε αυτούς τους οποίους χρειαζόμαστε αλλά και για την κοινωνική ασφάλιση έχουμε τόσο διαφορετικά συστήματα στις διάφορες χώρες δεν συμφωνούν ήδη μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως θα ικανοποιήσουμε λοιπόν τους εργαζόμενους από τρίτες χώρες. Θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο το θέμα. Θεωρώ ότι ο συμβιβασμός είναι τώρα καλός. Θα πρέπει να τον υπερψηφίσουμε γιατί έτσι θα έχουμε τουλάχιστον μία βάση. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα η κυρία Φλότρ για ένα λεπτό. Πρέπει να ομολογήσουμε πως είναι παράδοξο να ξεκινάμε μια οδηγία η οποία έχει ως στόχο να εγγυηθεί ένα νομικό πλαίσιο ε, πρόσβαση στα ίσα δικαιώματα για όλους τους εργαζόμενους από έναν μακρύ κατάλογο αποκλεισμού διαφόρων κατηγοριών εργαζομένων αυτή την οδηγία. Και αυτό παίρνει ξαφνικά τη μορφή μιας οικοδόμησης ε, ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας ως ένα μιλφέγγι όπου κάθε κατηγορία εργαζόμενου θα έβρισκε θέση ανάλογα με την εξειδίκευσή του κλπ. Άρα είμαστε μακρά από μια οριζόντια αντιμετώπιση του προβλήματος. Νομίζω ότι δεν έχουν καταλάβει οι Ευρωπαίοι υπεύθυνοι ότι εάν πετύχουμε αυτά τα οποία ζητάμε, τότε θα υπάρχουν ωφέλη και για τους μετανάστες, αλλά και για τις κοινωνίες υποδοχής και για τις κοινωνίες προέλευσης. Όπως το δείχνει μια μελέτη του London School of Economics, ότι αναφέρει ότι η νομιμοποίηση 600.000 παρανόμων στην Αγγλία που δεν θα έχουν δικαίωμα σε αυτήν την ενία άδεια θα ε, επιφέρει 3 δισεκατομμύρια λιβρών στην, ε, στα ταμεία της Μεγάλης Βρετανίας. Με συγχωρείτε τέλειος ο χρόνος σας και τώρα έχει ο κύριος Σογκόρ για δύο λεφτά. Θα ήθελα να πω ότι στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οικονομική μετανάστευση είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα και ω εκ τούτου χρειάζεται να έχουμε μια προσέγγιση διτή. Αφενός θα πρέπει να διαπιστώσουμε ότι το φαινόμενο αυτό ανταποκρίνεται σε μια οικονομική ανάγκη. Οι δημογραφικές τάσει που υπερισχύουν στην αγορά εργασία σημαίνει ότι στην Ευρωπαϊκή Κοινωνία απαιτούνται ε, μετανάστες εργαζόμενοι. Επιθυμούμε λοιπόν αυτή η μετανάστες να γίνεται σε ένα νόμιμο πλαίσιο και μπορούμε να ελέγχουμε τις απαραίτητες προϋποθέσεις και ο εργαζόμενος να αισθάνεται ότι εντάσσεται σε ένα νομικό πλαίσιο το οποίο δεν μπορεί να επιτρέπει την παράκαμψη αυτού του ε, νομικού πλαίσιου. Χρειάζεται λοιπόν να υπάρχει ένα κοινό ε, κατόφλη, δηλαδή σε ό,τι φορά την πρόσβαση σε δικαιώματα τόσο των ε, εργαζομένων υπηκών όσο και των υπηκών τρίτων χωρών. Ε, θα ήθελα να αναφερθώ στην πολιτιστική διάσταση. Διαπιστώνουμε ότι στα κράτη-μέλη υπάρχει μια σημαντική ένταση που προκαλείται με τους μετανάστες αυτούς. Θεωρώ ότι το να εξασφαλίσουμε αυτό το κοινό κατόφλι δεν μπορούμε να το πετύχουμε μέσω απογορεύσεων. Θα πρέπει να υπάρχει μια προσέγγιση λοιπόν ε, πιο ε, διαβαθμισμένη. Οι μετανάστες ε, θέλουν όχι μόνο να εργάζονται, αλλά θέλουν και να, δουλέψουν, να δημιουργήσουν οικογένειες, να ανατρέψουν τα τέκνα τους και να συμμετάσχουν στις κοινωνίες μας. Είναι ευρώ ότι επίλυση του προβλήματος μέσω της εργασίας θα οδηγήσει σε δημογραφική ανισορροπία δεν μπορούμε να αποκλείσουμε παράλληλα και τον πολιτιστικό ε, ζήτημα. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει αμοιβαία αναγνώριση, ανοχή αλλά και αλληλεγγύη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σκοφεράτη. Έχει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πιστεύω πως η λύση την οποία συζητάμε είναι μια λύση εσφαλμένη, βαθιά άδικη απέναντι σε πολλά αδύναμα άτομα, αλλά και νομίζω πως ε, μας πλήττει διότι εξάλλου αναφέρθηκε και από άλλους η αντίθεση η οποία υπάρχει ανάμεσα στο να συζητάμε μια ενία άδεια και να ξεκινήσουμε από εξαιρέσεις ε, και έναν κατάλογο εξαιρέσεων. Ε, αποκλεισμό των εποχιακών, των προσφύγων και των ε, ε, μετατεθειμένων ε, δημιουργεί ανισότητα τόσο στον τομέα της εργασίας όσο και στον τομέα των υπηκοτήτων. Εδώ δεν βρισκόμαστε μόνο απέναντι σε μια λύση η οποία μπορεί να οδηγήσει σε dumping διότι το κόστος θα είναι διαφορετικό ανάλογα με την χώρα αλλά θα υπάρχουν διακρίσεις ανάμεσα στους πολίτες. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να συζητήσει Επίσης το ζήτημα των σχέσεων με τους ε, εποχιακούς εργαζομένους. Κύριε Επίτροπε, δεν είναι πρόκειται μόνο για αλλοδαπούς, είναι και Ευρωπαίοι εποχιακά εργαζόμενοι. Αν οι μέθοδοι μας αποδογήσουν σε διακρίσεις και διακριτική μεταχείριση, τότε θα υπάρχει μια υποβάθμιση των ε, συνθηκών εργασία από τι επιχειρήσει, ό,τι φορά τη χρησιμοποίηση των ατόμων. Σε αφορά τώρα του αποσπασμένου, ε, αντιλαμβάνεστε τι θα συμβεί στι μεγάλε πολυεθνικέ, εάν ε, μπορούν να λαμβάνουν πλεονεκτήματα για πρόσωπα τα οποία θα έρχονται να εργαστούν σε εμά, αλλά θα προσλαμβάνονται με συνθήκες που ισχύουν στη χώρα προέλευσης. Είναι μια κατάσταση πρωτοφανής αλλά και καταστροφική. Όχι μόνο θα έχουμε το ντάπινγκ στην καθημερινότητα αλλά και η διαφορά ανάμεσα στους πολίτες που θα δημιουργηθεί που η Ευρώπη ποτέ δεν είχε στην ιστορία τους ακόμα και την πλέον πρόσφατη. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι θεμελιώδης η ενότητα και ως εκ τούτου το νομοθέτημα θα πρέπει ριζικά να τροποποιηθεί. Ευχαριστώ τώρα ο κύριος Κοέλιο για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Επίτροπε κυρίες και κύριοι. Ας είμαστε σαφείς. Είμαστε ενώπιον μιας ε, συμφωνίας που μας ικανοποιεί. Όχι. Σαφέστατα όχι. Πολλοί από εμάς θα θέλαμε να είχαμε πάει πιο μακριά. Πρόκειται όμως για ένα βήμα προς την ορθή κατεύθυνση για δύο κυρίως λόγους. Πρώτον, διότι δημιουργούμε ένα καινούργιο μέσο ε, που θα ωφελήσει τους υπηκόους τρίτων χωρών που θέλουν να στεύσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζοντάς τους μια σειρά δικαιωμάτων. Δεύτερον, όπως είπε και η Βερόνικ Ματιέ, ε, στέλνουμε και ένα πολιτικό μήνυμα ε, που αντιτίθεται με την Ευρώπη της καταστολής, την Ευρώπη φρούριο και οχυρό. Ε, θέλουμε μεταναστευτικέ πολιτικέ ευέλικτε για να προσπίσουμε τα συμφέροντα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνώ με την κυρία Ματιέ ότι χρειάζεται ε, να καταλήξουμε επιγόντω ε, σε συμφωνία με το Συμβούλιο. Η Σοφή Ιντβέλτ λέει βέβαια ότι πολλά κράτη-μέλη δεν επιθυμούν κοινή μεταναστευτική πολιτική, αλλά γι' αυτό ακριβώ το λόγο είναι σημαντικό να κάνουμε αυτό το πρώτο βήμα. Α είμαστε σαφεί. Η καταρρύξη των εσωτερικών συνόρων μεταξύ των κρατών μελών κατέστησε απαραίτητη την εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών σε ό,τι αφορά την ε, εισδοχή και την διαμονή υπηκών τρίτων χωρών προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμεταχείρισή τους με συγκρίσιμες υποχρεώσεις και δικαιώματα. Και πιστεύω ότι με την δημιουργία αυτής της διαδικασίας νέας άδεια και την χορήγηση τέτοιου είδους αδειών θα γίνουμε πιο αποτελεσματικοί και οι εργοδότες και οι μεταναστές εργαζόμενοι και ταυτόχρονα θα μας επιτρέψει να ελέγχουμε πιο εύκολα ε, την ε, εργασία τους και την διαμονή τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η επόμενη ομιλήτρια είναι η κυρία Σερακιάνη για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σήμερα η πρόσβαση στην ε, εργασία ρυθμίζεται μόνο για ορισμένες κατηγορίες πολιτών τρίτων χωρών. Δεν ε, απολαύουν όλοι την ίση μεταχείριση σε ό,τι φορά την πρόσβαση στην εργασία. Σε αυτό το πλαίσιο η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται να δράσει προκειμένου να εξασφαλίσει την ισότιμη μεταχείριση των νομίμως διαμενόντων όσο και των όσων έχουν το καθεστώς διεθνούς προστασίας ή πρόσφυγες σύμφωνα με την οδηγία του 83 του 2004. Πρέπει να αποφύγουμε να υπάρχουν ε, συνεχή αιτήματα για εποχιακούς επειδή πληρώνονται λιγότερο ή και κοστίζουν γενικά λιγότερο από έναν Ευρωπαίο που κάνει την ίδια δουλειά. Θα πρέπει να αποφύγουμε τον κίνδυνο πολλές πολυεθνικές να μεταφέρουν τας, ε, τις, ε, τα γραφεία τους σε χώρες της Βορειοαφρικής. Ε, θα πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε την απαραίτητη και την ίση ε, μεταχείριση, συνθήκες εργασία, ε, κοινωνική πρόνοια κλπ. Θεωρώ λοιπόν ότι οι πρόσφυγες, οι ανεξάρτητοι επιχειρηματίε και οι τα αποσπασμένοι να ενταχθούν σε αυτήν την οδηγία. Αν κάνουμε διακρίσεις θα οδηγηθούμε σε με έναν ιδιαίτερα ολίστερο δρόμο. Ευχαριστώ. Good evening, my dear colleagues. I've just arrived from... Ε, καλησπέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Μόλις έφτασα από τη Φραγκφούρτη ε, και υπήρχε μεγάλη συμφόρηση στο δρόμο. Ελπίζω ότι δεν θα κάνω λάθη εις ε, την διεξαγωγή της Προεδρίας της συνεδρίασης και θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Ελίζα Γιακονσάρη για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, εδώ και αιώνες η Ευρώπη γνώρισε το φαινόμενο της ε, απομάκρυνσης, εγκατάλειψης ε, λόγω ε, πολλών και διαφόρων αιτιών. Ε, τώρα όμως χρειάζεται να δείξουμε κατανόηση για τους ε, πολίτες τρίτος χωρών που έρχονται από τις χώρες τους. Χρειάζεται λοιπόν να ε, βρούμε έναν τρόπο για την επίλυση του προβλήματος αυτού. Νομίζω πως η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι σωστή. αυτή η προσέγγιση η τομεακή θα πρέπει να προσφέρει εγγύηση στους εργαζόμενους αλλά έχουμε οδηγηθεί δυστυχώς σε μια απαράδεκτη κατάσταση. Ποιοι πολιτική μετανάστευση. Υπάρχουν πρόσωπα που φτάνουν με μπλε υπάρχουν εποχιακοί, υπάρχουν ε, πρόσωπα τα οποία είναι ενδοεπιχειρησιακά ε, αποσπασμένα γιατί η Κομισιόν δεν κατορθώνει να εφαρμόσει τους ίδιους κανόνες για όλους τους ε, εργαζομένους. Ε, σε διάφορες παρεμβάσεις ακούσαμε πως ορισμένες κατηγορίες μεταναστών παραμένουν εκτός του πλαισίου του νομοθετικού. Αυτό είναι απαράδεκτο. Πρέπει να υπάρχει ίση μεταχείριση και αντιμετώπιση όλων των μεταναστών. Δεν πρέπει λοιπόν να επιτρέπουμε άλλα να γίνονται δεκτοί και άλλοι να αποκλείονται. Η ομάδα μας, η ομάδα των σοσιαλιστών, έχει υποβάλει κάποιες τροποποιήσεις και ελπίζω αύριο κατά τη διάρκεια των ψηφοφοριών να γίνουν δεκτές. Το κείμενο λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Χρειάζεται οι διατάξεις νομοθετικέ, νομοθετικές να είναι ισότιμες για όλους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Εύελιν Ρέινιε για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Η ιδέα του One Stop Shop είναι πολύ καλή, αλλά ε, για ορισμένες χώρες όπως η δικιά μου, η Αυστρία, μία χώρα όπου η άδεια παραμονής δίδεται από την υπηρεσία αλλοδαπών, ενώ εργασίας από την ε, ε, υπηρεσία εργασίας που υπόκειται στον έλεγχο των κοινωνικών εταίρων. Άρα και οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει να συμμετάσχουν σε αυτή τη διεργασία και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και η Εκκλησία δεν έχουν εμπλακεί αρκετά. Θεωρώ ότι είναι ένα σύνολο και δεν μου αρέσει αυτή ο κατακαιρματισμός του πακέτου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ε, θεωρώ ότι πρόκειται για κοινωνικό υποβιβασμό. Θέλω να κάνω μία παρατήρηση όσον αφορά το επιπρόσθετο έγγραφο, διότι ε, ήδη στην επιταγή όλα μπορούν να περιληφθούν. Άρα το έγγραφο αυτό πρέπει να επιτρέπει καλύτερο έλεγχο για να υπάρχει μεγαλύτερη προστασία των εργαζομένων και να αποφευθεί μία στρέβλωση του ανταγωνισμού υπέρ των επιχειρήσεων οι οποίοι θέλουν να πλουτίσουν βάσει παρανόμων εργαζομένων. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα δίνω τον ε, λόγο ε, εις ε, τη διαδικασία Catch the Eye και πρώτα Η κυρία Ουμαν Ρόιτερ έχει το λόγο. Πρόεδρε, είχα ε, ζητήσει δύο-τρεις φορές το λόγο προηγουμένως. Ε, έχω την εντύπωση σε αυτή τη συζήτηση ότι, ε, δεν έχουμε ασχοληθεί με, το, την κοινωνική πτυχή του θέματος αυτού. Εγώ έχω υποβάλει μια τροπολογία που έχει ως στόχο να χορηγήσει την ε, ίση μεταχείριση, την ίδια μεταχείριση σε όλα τα άτομα που θα φτάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση, αυτή ε, με βάση αυτήν την ενιαία άδεια. Ε, πουθενά δεν αναφέρεται ότι δεν εγγυόμαστε κάτι τέτοιο. Διάβασα τα άρθρα ένα προς ένα και έχω την εντύπωση ότι δημιουργούμε ένα λαθασμένο σύστημα. Ε, οι εποχιακοί εργαζόμενοι ε, δεν καλύπτονται αυτή τη στιγμή. Ε, είναι δυνατόν να δημιουργηθεί επίσης μια εταιρεία σε μια τρίτη χώρα από κάποιους Ευρωπαίους και να αποστέλουν μετά από εκεί επιχειρησιακά εργαζόμενους και να εργάζονται στις χώρες μας. Τώρα ερχόμαστε σε τη διαδικασία Catch the Eye και πρώτος ο μιλητής είναι ο κύριος Μαρινέσκου. Κύριε Πρόεδρε, εκτός μικροφώνου ο κύριος Σέρκας. Mulțumesc, domnule președinte Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η ενία άδεια θα διευκολύνει τι διοικητικέ διαδικασίε και θα διευκολύνει και την ανταλλαγή δεδομένων στο πλαίσιο τη οικονομική μετανάστευση. Θεωρώ λοιπόν πω αυτή η νομοθήκη πρόταση επιλύει όμω το πρόβλημα κατά το ίμιση διότι έχουμε ήδη άτομα τα οποία έχουν γίνει αποδεκτά στην επικράτηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν καλύπτουν ε, τις δύο απαντές προϋποθέσεις ε, που αφορά τους εποχιακά εργαζόμενους και τους ε, ενδοεπιχειρησιακά μετατιθέμενους. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εδώ φροντίζουμε να ρυθμίσουμε τα δικαιώματα των πολιτών τρίτων χωρών, αλλά δεν έχουμε μια ελεύθερη αγορά ούτε ακόμα, ούτε καν για τους Ευρωπαίους πολίτες. Ευχαριστώ και βουλευτά. Κυρία λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε συζητήσει πολύ για ισότητα δικαιωμάτων, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει ε, επίσης είναι ε, και ε, η διεκπαιρέωση και τα βραχυπρόθεσμα αλλά και τα μακροπρόθεσμα μέτρα διότι γνωρίζουμε ε, που κατέληξε η οδηγία σχετικά με την παροχή υπηρεσιών και τι ε, σημασία της ε, δόθη απερίθμησε το σύστημα το οποίο χειροτέρεψε και δεν βελτιώθηκε εδώ λοιπόν μας απειλεί μία κοινωνική καταστροφή για διάφορους κλάδους οι οποίοι θα χρειαστεί να αναλάβουν εργασία και αυτό θα συμπιέσει προς τα κάτω τους μισθούς. Δεν ξέρω ποιες είναι οι απόψεις των άλλων πολιτικών ομάδων αλλά εμείς δεν μπορούμε να στηρίξουμε κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν τέτοιες εξαιρέσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε κοινωνικές διαταραχές. Η κυρία Αλφάνο έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, ο ΙΕ ε, ενέκρινε την ε, οδηγία για τα μετανάστες εργαζόμενους για τις οικογένειές τους και αποτελεί ένα από τα βασικά θεμέλια εδώ και 20 ε, χρόνια. Μετά από 20 χρόνια όμως κανένα από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ε, επικύρωσε αυτή τη σύμβαση. Τα αναγνώριση των δικαιωμάτων των πολιτών τρίτων χωρών που ε, διαμένουν και εργάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει μια Ευρώπη η οποία οποία προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γι' αυτό λοιπόν προτείνω στους συναδέλφους να ε, υπερψηφίσουν την ε, τροπολογία υπερθυμών 16 και την ε, αίτημα το οποίο έχουν καρθέσει με την Κέλλαρ όπου ζητάμε την επικύρωση της σύμβασης του ΟΗΕ για τους εργαζόμενους. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει στήσει η κυρία Ρέιδο για ένα λεπτό. Η πρόταση αυτή κάνει λόγο για πολλές και διαφορετικές καταστάσεις συμπεριλαμβανομένων μεταναστών από τρίτες χώρες, εποχιακών εργαζομένων και ε, άλλων κατηγοριών. Όμως ε, αυτό που προσπαθούμε στην πράξη είναι να ε, νομοποιήσουμε το κοινωνικό dumping και να ενισχύσουμε την εργασιακή ανασφάλεια αυξάνοντας ε, τις ε, ανισότητες. Γι' αυτό το λόγο λέμε ότι αυτή η πρόταση οδηγίας δεν είναι δυνατόν να γίνει δεκτή. Χρειάζεται να βελτιώσουμε τα δικαιώματα των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι που χρειάζεται όποιοι και αν είναι αυτοί οι εργαζόμενοι, ε, μερικής απασχόλησης, εποχιακοί, μετανάστες κλπ. Πρέπει να αναγνωρίσουμε τα δικαιώματά τους μέσω μιας τέτοιας οδηγίας, συμπεριλαμβάνοντας και τη Διεθνή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων όλων των ε, εργαζομένων και μεταναστών και των οικογενειών τους. Ε, είναι ώρα η Κομισιόν να υποβάλει μια τέτοιου πρόταση, η οποία θα εγκριθεί και θα υιοθεθεί από τα κράτη-μέλη και, να, και τη σύμβαση να επικυρωθεί επίση. Ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Γιάρος Τραχμόσκα έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το θέμα της ε, μετανάστευσης είναι γνωστό στις πιο πλούσιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σαν συνηθισμένο φαινόμενο και εκτός από τους νόμιμους υπάρχουν και οι παράνομοι μετανάστες οι οποίοι υφίστανται ε, εκμετάλλευση και διακρίσεις. Η προσπάθεια να οργανωθεί το θέμα και να εφαρμοστούν νέοι κανόνες, κάτι το οποίο ε, θέτει αυτή η οδηγία είναι ένα θετικό στοιχείο. Βεβαίως αυτό που είναι σημαντικό είναι οι μετανάστες να δεχθούν αυτούς τους κανόνες γνωρίζοντας ότι δεν πρόκειται να λυθούν όλα τα προβλήματά τους. Ε, υπάρχουν και θετικά στοιχεία τα οποία αντιμετωπίζουμε και γι' αυτό η πρόταση ε, για τη νέα οδηγία δεν μπορεί να θεωρηθεί σαν ένα θετικό βήμα. Ευχαριστώ και το λόγο έχει τώρα ο Σον Κέλλη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Έχουμε στην Ιρλανδία ένα ρητό. Και αν μπορούμε να εφαρμόσουμε ε, το ρητό κάπου είναι εδώ διότι ο εισηγητής έχει κάνει ε, μια εξαιρετική εργασία και ε, προσπαθεί να επιβάλλει ειρήνη και ευημερία σε ολόκληρο την Ευρωπαϊκή Ένωση και στον κόσμο. Επειδή λοιπόν ο κόσμος πρέπει να προστατεύσει τις υποανάπτυξη χώρες, θα πρέπει και οι, υπήκοοι των τρίτων χωρών να την χάνουν του ίδιου σεβασμού τον οποίο επιζητούμε για τους δικούς μας. Τίποτα όμως δεν είναι τέλειο και γι' αυτό θέλω να σας πω ότι θα στηρίξω τον εισηγητή. Ευχαριστώ και με κάποια καθυστέρηση επιτέλους δίνει το λόγο στον κύριο Σέρκας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν θέλω να ξεκινήσω συζήτηση με τη συνάδελφο Αμενρόιτεν, αλλά για να διευκρινίσω κάποια ζητήματα. Δεν υπήρχε καμία συζήτηση και καμία αφισβήτηση των εργασιών της. Εγώ προσωπικά να δηλώσω ότι έκανε εξαιρετική δουλειά στην Επιτροπή Απασχόληση. Αλλά αν η κυρία Νόρμεν ε, ο Μενρόιτερ είπε ότι καταθέτει τροπολογίες οι οποίες βελτιώνουν την έκθεση, θα έλεγα πως όχι. Ε, έχει υπογράψει τις ε, τροπολογίες τις οποίες το Κοινοβούλιο δεν, το Συμβούλιο συγγνώμη, δεν μπόρεσε να δεχθεί στο κείμενο. Μιλάμε τώρα για το κείμενο του Συμβουλίου και σε ό,τι αφορά την απόσπαση η θέση του Συμβουλίου ήταν πολύ διαφορετική από το κείμενο της Κομισιόν. Αλλά εμείς δεχόμαστε την πρόταση της Κομισιόν. Αλλά το κείμενο του Συμβουλίου λέει ότι όλοι οι μετατιθέμενοι, συμπεριλαμβανόμενοι και αυτών της οδηγίας εντέξει αποκλείονται από τη συγκεκριμένη οδηγία. Δεν πρόκειται για ισότητα, αλλά για ε, ανισότητα. Ε, ε, εγώ πω ότι είναι μια εξαίρετη βουλευτής η κυρία Ομενρόιτερ, εργάστηκε άψογα, αλλά τελικά λέει τα πράγματα με το Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Μην ε, εκνευρίζεστε κυρία Όμιν Ρόιτεν, δεν μπορώ να σας ε, ξαναδώσω το λόγο, διότι ε, φτάσαμε στο τέλος της συζητήσεως επί του θέματος και σας ζητώ τώρα να ακούσετε την κυρία Μέλστρομ που λαμβάνει το λόγο ξενόματος της Κομισιόν. Κυρία Επίτροπε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όντως ήταν πολύ προβληματική συζήτηση. Σε ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογή, δεν είναι μυστικό ότι η Κομισιόν θέλει να έχει μια σφαιρική προσέγγιση. Φυσικά. Ε, ο προκάτοχός μου το πρότεινε πριν από πολλά χρόνια, αλλά ήταν κάτι το οποίο δεν ε, επιτεύχθηκε. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε αυτή την κλαδική προσέγγιση, αλλά με αυτό θα πρέπει να προχωρήσουμε. Είναι απαραίτητο διότι έχουμε τους εργαζόμενους επικός τρίτων χωρών που συνεισφέρουν σημαντικά στην οικονομία μας και θέλουμε να τους προστατεύσουμε. Τούτου λεχθέντος να αναφερθώ σε κάποιες από τις απόψεις που εκφράστηκαν. Να τονίσω ότι η οδηγία ε, αναφέρεται στην αρχή της ίση μεταχείρισης σε όλες τις θέσεις εργασίας συμπεριλαμβανομένων και των συνθηκών εργασίας και της, ε, των αμοιβών. Δεν δημιουργεί διακρίσεις. Όταν εγκριθεί θεωρώ ότι θα ήταν ένα πολύ σημαντικό εργαλείο προκειμένου να, να αγωνιστούμε για την κατά του κοινωνικού ντάμπινγκ. Εμεί θέλουμε να προστατεύσουμε αυτά τα πρόσωπα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τι κατηγορίε εργαζομένων, δεν έχουν συμπεριληφθεί στην πρόταση αυτή, όπω οι εποχιακά εργαζόμενοι και οι ενδοπιχειρησιακά μετεκτέμενοι. Θέλουμε να του προστατεύσουμε και αυτού. Γι' αυτό το λόγο, πριν από το φέρο, η Κομισιόν πρότεινε δύο διαφορετικά εργαλεία για τις ε, για τους ενδοπιχειρησιακά μεταθυμένους και για τους εποχιακούς και έχουν ως στόχο να τους προστατεύσουμε και οι συγκητές και οι συγκητές και οι αρμόδιες κοινοβουλικές τροπές όταν εξετάσουν το ζήτημα θα δουν ότι και αυτοί προστατεύονται από τις προτάσεις της Κομισιόν. Επίσης κατανοώ ότι οι ορισμένε πολιτικές ομάδες θα ήθελαν να ε, έχουν συμπεριληφθεί να έχουν συμπεριφθεί και η αποσπασμένη. Η οδηγία την οποία συζητάμε σήμερα ε, επιθυμεί να αποφευχθούν οι διακρίσεις και όχι τη δημιουργία νέων. Γι' αυτό λοιπόν ας εξετάσουμε το ζήτημα των ε, αποσπασμένων διαφορετικά. Η Κομισιόν θα κάνει μια μελέτη αντικτύπου ε, επί του θέματος αυτού. Προβλέπεται μια αναθεώρηση της οδηγίας για τους μετατιθέμενους και σε ό,τι αφορά τώρα το θέμα των πινάκων αντιστοιχία, ναι, η Κομισιόν ε, συμμερίζεται αυτή την άποψη, όχι μόνο σε αυτή την οδηγία, θα ήταν και θα είναι ένα σημαντικό εργαλείο για το θέμα της βέλτιστης νομοθεσίας και τη καλύτερη διαφάνεια στα κράτη-μέλη κατά την εφαρμογή των ε, οδηγιών. Θα είναι καλό για εσά, για τα εθνικά κοινοβούλια, για εμά και για του πολίτε. Και συνεχίζουμε να το επαναλαμβάνουμε προ το Συμβούλιο ότι κάτι τέτοιο θα διευκόλυνε την Κομισιόν στο να υποβάλει μια δήλωση. Πάντως ε, ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να ε, βρούμε μια λύση, όχι εντός της αύριο φυσικά. Τώρα, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για τη συζήτηση, ευχαριστώ για τη σκληρή δουλειά που πολλοί εξημών έκαναν, ο κύριος Έργας, κυρία Ματιώ και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να πετύχουμε συμφωνία και να υπάρξει θετική ε, ψήφιση, ψηφοφορία αύριο, η υπερψήφιση. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Και τώρα να δώσω το λόγο στην Βερονίκ Ματιού, η Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Δεν θέλω παρά μόνο να συμφωνήσω μαζί σας διότι απαντήσατε θαυμάσια στους 23 συναδέλφους οι οποίοι επενέβησαν σχετικά με το κείμενό μας του κυρίου Σέρκας και το δικό μου. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εισηγητές επί του θέματος αυτού και για τις πολιτικές ομάδες όλες με τις οποίες είχαμε με μεγάλο διάλογο και πολύ καλή συνεργασία συνεργασία καθόλου το έτος διότι η συνεργασία αυτή σε ένα έτος άρχισε στην αρχή του χρόνου και τελειώνει με τη Βελγική Προεδρία ευχαριστώ και την κυρία Μάλστρομ η οποία εισάκουσε τα σχόλιά μας και τις υπηρεσίες οι οποίες μας πρόσεξαν πολύ ε, και στο Συμβούλιο και θέλω να ευχαριστήσω επιπλέον όλους τους συναδέλφους που επενέβησαν απόψε. Θα ήθελα να πω ότι ουσιαστικά αύριο θα έχουμε την ψηφοφορία σε πρώτη ανάγνωση και πρόκειται για ένα συμβιβασμό. Ο συμβιβασμός βέβαια ποτέ δεν είναι πλήρως ικανοποιητικός και αν υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι ζητούν να καθησυχαστούν ίσως τα σχόλιά σας τους καθησυχάσουν η Ελέν Φλότερ που είπε προηγουμένως ότι ξεκινά ένα κείμενο εκθέσεως με εξαιρέσεις σας υπενθυμίζω ότι όλοι οι εργαζόμενοι οι οποίοι, στους οποίους αναφέρονται οι εξαιρέσεις καλύπτονται από άλλες ε, από άλλα θέματα και γι' αυτό το κείμενο το οποίο επιτύχαμε και καταρτήσαμε με όλους τους ηγητές και θα υποβάλουμε αύριο ή στους συναδέλφους θα είναι ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός για τους εργαζόμενους από τρίτες χώρες ευχαριστώ. Σας εύχομαι καλή επιτυχία και έτσι ολοκληρώνεται η συζήτηση. Αύριο θα ψηφίσουμε και προχωρούμε τώρα